Herr Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Ich erkläre die am 24. Η σύνοδος που διακόπη στις 24 Νοεμβρίου 2016 αναλαμβάνεται. τα πρακτικά και τα κείμενα της 24 η Νοεμβρίου. Τα έχετε στη διάθεσή σας, δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει.